Νότιο Σουδάν τώρα, μεταξύ ε, των θεμάτων είναι και το θέμα των απαγωγών παιδιών. Θα δώσω το λόγο στην ε, πρώτη εισηγήτρια, την κυρία Τζούντιτ Σαρτζεντίνη. Ένα λεπτό, έχει το λόγο. Ε, Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε καμιά ιδιαίτερη εισαγωγή εδώ. Τα έχει εξηγήσει αυτά, νομίζω επανειλημμένα τα έχουμε συζητήσει στο Κοινοβούλιο. Δυστυχώς τα προβλήματα στη χώρα αυτή το πληρώνουν οι πληθυσμοί και πρόσφατα ε, έπεσαν θύματα απαγωγής 89 παιδιά, μπορεί και περισσότερα στο νότιο Σουδάν. Παιδιά από 12 ετών και άνω αγόρια από 12 ετών και άνω που καλούνται να υπηρετήσουν σαν στρατιώτες ε, σε κάποιο από τα ε, αντιμαχόμενα συμφέροντα. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα βιβλίο που είχε βγει στην ουσία το 2006 το οποίο λέγει ακριβώς τι είχε ζήσει ένας νέος ο οποίος είχε πέσει θύμα απαγωγής, ο οποίος το έσκασε, ε, διέσχισε μόνος του και κατέληξε σε ένα στρατόπεδο προσφύγων. Πρέπει τα παιδιά αυτά να απελευθερωθούν το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ ο κύριος Γέζεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που βλέπω ότι συμφωνούμε σε ένα τέτοιο θέμα. Αυτό σημαίνει ότι συνειδητοποιούμε πλήρως τις καταστροφές αυτές στο Νότιο Σουδάν. 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένοι, 500.000 έφυγαν σε γειτονικέ χώρες, 2.000 παιδιά αναγκάστηκαν να πάρουν τα όπλα και φυσικά χιλιάδες θύματα, βιασμοί, ε, παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα διατροφικά, και γι' αυτό το Κοινοβούλιο δικαιολογημένα ζητά από τη διεθνή κοινότητα να οργανώσει μια συνάντηση δωρητριών χωρών για τον Νότιο Σουδάν έτσι ώστε να ε, πληρωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Εγώ συμφωνώ με αυτά τα οποία λέμε στο κείμενο, ακούω αυτά τα οποία μας ε, λένε και μας ενημερώνουν ε, οι τοπικοί πληθυσμοί ε, δυστυχώς τα στοιχεία μιας ευρυτά της καταστροφής έχουν πλέον αρχίσει να συγκεντρώνονται. Ε, θα πρέπει να υπάρξει μια ομάδα επαφής ε, για τον Νότιο Σουδάν. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε μια συνεκτικότητα στον τρόπο παρέμβασής μας. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ζετνάνσκα. Ευχαριστώ. Στους πολέμους πρώτα θύματα είναι πάντα τα παιδιά. Χιλιάδες είναι τα παιδιά που έχουν ε, αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σχολεία τους, αλλά και πολλά, ακόμα τώρα τελευταία το Φεβρουάριο, που απάγονται για να μετατραπούν σε στρατιώτες στο Σουδάν. 89 μόνο το Φεβρουάριο. Παίρνουν μια σύντομη εκπαίδευση και μετά τα ρίχνουν στον πόλεμο. Παιδιά τα οποία θα στιγματίσει αυτή η εμπειρία για όλη τη ζωή. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να εκφράσουμε όλοι την ικανοποίησή μας για τις κυρώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατά εκείνων των ηγετών του Νότιου Σουδάν που θέλουν να παρεμποδίσουν την ειρηνευτική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοράου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω οποιοδήποτε σχόλιο για, για το απάνθρωπο, για το φρικαλαίο των όσων συμβαίνουν στο Νότιο Σουδάν είναι περιττό. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα να τα απαριθμούμε και να λέμε πόσο αποτρόπαιο είναι αυτό που συμβαίνει σε αυτά τα παιδιά στρατιώτες, αλλά και στα κορίτσια τα οποία βιάζονται, ε, απάγονται και τις χρησιμοποιούν ως δούλες ή σκλάβες και κατευθύνονται μετά στην αγορά πορνείας. Στο νότιο Σουδάν έχουμε ένα από τα νεότερα κράτη παγκοσμίω και βεβαίως πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε ότι από τη στιγμή που δημιουργήθηκε βρίσκεται σε μια κατάσταση εμφύλιας σύγκρουσης, διαρκείας. Οπότε τι λόγο έχουμε να διατηρούμε το κράτος αυτό σε αυτή την κατάσταση, ποιος έχει οικονομικά συμφέροντα για να ε, διατηρεί την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται και να ε, συνεχίζονται αυτές οι απάνθρωπες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Εντάξει, των συντακτών η κυρία Χιμένες Μπεσερίλ Μπαρίο. Μπαρίο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Νότιο Σουδάν είναι μία από τις χειρότερες στον κόσμο. Η ειρήνη δεν έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες από το 2011 που έγινε ανεξάρτητη η χώρα ξεκίνησε ένας εμφύλιος πόλεμος με καταστροφικές συνέπειες για τα παιδιά, για τα κορίτσια τα οποία πέφτουν θύματα σεξουαλικής βίας και φυσικά υπάρχει και το θέμα των παιδιών στρατιωτών. Οι αριθμοί είναι ιδιαίτερα απογοητευτικοί. Υπάρχουν παιδιά τα οποία συλλαμβάνονται, βιάζονται, φυλακίζονται. Το πρόγραμμα δράσης ε, δυστυχώς έχει το πρόγραμμα το ειρηνευτικό το οποίο είχε εφαρμοστεί έχει παραβιαστεί και συνεχίζεται η εκμετάλλευση των παιδιών σαν στρατιώτες που δεν μπορούμε να το παραδεχτούμε. Νομίζω ότι ε, δεν μπορούμε να αφήσουμε τέτοιου είδους βαρβαρότητα και πρέπει να βρούμε κάποια λύση σε αυτήν την σοβαρότατη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λίντια Σένρα Ροντρίγκε μεταξύ των συντακτών. Ε, για ένα λεπτό πάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταδικάσουμε τέτοιου είδους βία εις βάρος των παιδιών, των ε, κοριτσιών και των αγοριών Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και ε, επίσης ένα από τα προβλήματα αυτά είναι και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις διπλωματικές οδούς έτσι ώστε να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υπάρξει τέλος ε, στα, στα, παιδιά, στα, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά πρέπει να ανακτήσουν την παιδική τους ηλικία, πρέπει ε, να εκριζώσουμε επίσης και την φτώχεια έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα οικονομικής στήριξης να μπορούν να παράγουν τα τρόφιμα οι περιοχές αυτές για να ζήσουν τους τοπικούς πληθυσμούς. Ευχαριστούμε. μεταξύ των συντακτών ο κύριος Βάιντενχόλτσερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά πρέπει να συζητήσουμε την κατάσταση του Νότιου Σουδάν. Η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς. Καταστρέφονται κρατικές δομές. Επικρατεί κοινωνική εξαθλίωση. Λέγαμε τον Νοέμβριο πέρυσι ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση και τίποτα δεν έχει συμβεί. Έχει ακόμα επιδεινωθεί η κατάσταση. Είναι ακόμα πιο πολλοί οι πρόσφυγε έχουν φτάσει στους 5, 5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια, το 1 τέταρτο του πληθυσμού, αντιμετωπίζει το λοιμό. Επιπλέον αρχίζουν τώρα να χρησιμοποιούν και παιδιά ως στρατιώτες. Το μέλλον δηλαδή της χώρας κινδυνεύει από εξαφάνιση. Δεν πρέπει να σιωπούμε. Πρέπει να υψώσουμε το ανάστημα και τη φωνή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βάιντεν Χόλτσερ. Εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων τώρα, των πολιτικών ομάδων και δι του ΕΛΚ, ο κύριος Στίερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πριν από τέσσερα χρόνια περίπου ζήτησε το Νότιο Σιδάν και οι πολίτες του την ανεξαρτησία. Έκτοτε τα χαμένα αγόρια όπως ονομάζονται, παιδιά, μια γενιά ολόκληρη που είχαν υπηρετήσει ως παιδιά στρατιώτες, αποφάσισαν να γυρίσουν στη χώρα τους για να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον για αυτήν. Τα χαμένα αυτά αγόρια, αυτά που είχαν φύγει πρόσφυγες για να γλιτώσουν από τον πόλεμο, δυστυχώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νέα εμπόλεμη κατάσταση στη χώρα τους. Τον Ιανουάριο του 2013 ξέσπασαν βίες συγκρούσεις, εμφύλιες συγκρούσεις και αυτή η χαμένη παιδικότητα ήταν η μοίρα μιας ακόμη γενιάς παιδιών. Χιλιάδες είναι τα παιδιά στρατιώτες που χρησιμοποίησαν και οι δύο πλευρές της σύγκρουσης Πρόσφατα είδαμε και απαγωγές παιδιών στο Νότιο Σουδάν που μας υπενθυμίζουν αυτό το φαινόμενο. Εγώ υποστηρίζω τις κυρώσεις των ΗΕ προκειμένου να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να χρησιμοποιούν παιδιά ως στρατιώτες. Ευχαριστώ εκ μέρους της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών η κυρία Άννα Γκόμες, 1,5 λεπτό. Η απαγωγή και στατολόγηση παιδιών από τις ένοπλες δυνάμεις ε, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στο Νότιο Σουδάν είναι μια ένας πόλεμος που ξεκινά με, που κρατάει εδώ και ένα χρόνο με αποτυχημένες προσπάθειες ειρήνευσης με ιδιαίτερε ανθρωπιστικέ ανάγκε από την έναρξη αυτή τη σύγκρουση και στο κλίμα ατιμορρησία που η διεθνή κοινότητα δεν μπορεί να συνεχίσει να ανέχεται. Η ολοκλήρωση των ε, συνομιλιών για την ειρήνη έχουν οδηγηθεί σε παταγώδη αποτυχία και βασικά όλε οι δυνάμει τη περιοχή πρέπει να σταματήσουν να έχουν συμμετοχή στη σύγκρουση χωρί ε, μεροληπτική δράση και μόνο. Εδώ και ένα χρόνο προβλέπονται ε, μέτρα κατά των ηγετών που οδήγησαν σε μπλοκάρισμα τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Θα πρέπει να σταματήσει η διακίνηση όπλων στην περιοχή και να σταματήσουμε να αξιοποιούμε τα κέρδη από την πώληση πετρελαίου της περιοχής. Χρησιμοποιείται για σκοπούς πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να πιέσουν την Αφρικανική Ένωση να τοποθετηθεί και να δημοσιεύσει την έκθεση της Ανακριτικής Επιτροπής για το ε, τη εκταστική Μάλλον Επιτροπή για τον Νότιο Σουδάν. Θα πρέπει η ατιμορρησία ε, και η έλλειψη δικαιοσύνη και ο πόλεμο να λάβουν ένα τέρμα σε αυτή την περιοχή. Κάτω. Ευχαριστούμε. Εκ μέρου τη ΑΛΔΕ των Φιλελευθέρων η κυρία Γκρισμπέκ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, Ουσιαστικά είμαστε μάρτυρες τόσων ε, πολέμων ε, ανά τον κόσμο, ε, δημοκρατικών πολιτευμάτων που καταραίουν και οι πολίτες αναγκάζονται να μπουν ε, και να κρυφτούν στο καβούκι τους, ε, όπως το Νοτιού Σουδάν, όπου η χώρα είναι θέατρο ε, ενόπλων σειράξεων μεταξύ αδελφών, χιλιάδες παιδιά χάνουν τη ζωή τους, δολοφονούνται, απάγονται, βιάζονται, νεαρά κορίτσια γίνονται σκλάβες, εξαντραποδίζονται και τα παιδιά γίνονται στρατιώτες, είναι φρίκοι δεν αρκεί να εκφωνούμε ωραίε ομιλίε και να υπογράφουμε ένα ψήφισμα, αλλά πρέπει να δράσουμε. Δεν μπορεί να παραμένει αδρανή η διεθνή κοινότητα ενάντια μια τέτοια καταστροφή. Πρέπει να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσει και αμέσω να πάυσουν αυτέ οι βίε πράξει που είναι όνειδο για τη διεθνή κοινότητα και απαιτούν την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Madame ε, Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σον Κέλλη, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από δύο χρόνια, τρία χρόνια περίπου που πήρε την ανεξαρτησία του, προγνωρίστηκε την ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν, θυμάμαι να μιλάω εδώ πάλι στο Κοινοβούλιο με ελπίδα για την πρόοδο της νέας αυτής χώρας. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο όταν επικρατεί εμφύλιο πόλεμος σε μια χώρα, όπως τώρα στο Νότιο Σουδάν, δεν υπάρχει περίπτωση να προοδεύσει. Όταν φτάνουν να χρησιμοποιούν ακόμη και νεαρά παιδιά ως στρατιώτες. Όταν μπαίνουν στα σπίτια και τα σχολεία, βγάζουν τα γόρια από τις τάξεις τους ή από τα δωμάτια τους και ε, τους δίνουν στο χέρι ένα όπλο για να σκοτώσουν κάποιον άλλον. Δεν μπορούμε εμείς να μένουμε αμέτωχοι. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να θέσουμε ένα τέρμα στη βαρβαρότητα αυτή. Οι πόροι, τεράστιοι πόροι πετρελαϊκοί, πρέπει να αξιοποιηθούν για τη χώρα, για τον λαό της, για τα παιδιά της. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι τώρα πάμε στη δικασία Καρστιάη. Και δίνω το λόγο στον κύριο Νότι Μαριά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε το νότιο σουδάν είναι μια πλούσια περιοχή έχει τεράστιες πετρελαιοπαραγωγικές δυνατότητες και βεβαίως με το που απέκτησε την ανεξαρτησία του ήταν δεδομένο ότι ξένα συμφέροντα αξιοποιώντας τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις που υπήρχαν στην κοινωνία οδήγησαν την περιοχή αυτή σε ένα εμφύλιο πόλεμο. Τώρα πλέον έχουμε 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένους, έχουμε 500.000 πρόσφυγες σε γειτονικά κράτη, έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό στις συνεδριάσεις του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε μια ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή καθώς κινδυνεύουν πάνω από τέσσερα εκατομμύρια ψυχές. το νέο θέμα που υπάρχει είναι ότι τα παιδιά στρατολογούνται πλέον σε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο και μάλιστα γίνονται και απαγωγές παιδιών προκειμένου να υπάρξει βίαιη στρατολόγησή τους πρέπει να υπάρξει άμεση καταλυτική δράση της ευρωπαϊκής ένωσης στο θέμα αυτό για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την ανθρωπιστική κρίση. ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. do you accept blue card? Δέχεστε μια μπλε κάρτα από την κυρία Πέτυρ, παρακαλώ. παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Με συγκλονίζει η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν, καθώς καθημερινά γίνονται απαγωγές παιδιών που επιστρατεύονται ως στρατιώτες, αφού τα αφαιρούν από την ε, οικογένειά τους, τους δίνουν όπλο στο χέρι. Οι γυναίκες βιάζονται. Όσοι επιβιώνουν όμως από την κατάσταση αυτή και δυστυχώς λόγω της επιστημιστικής κρίσης και των πολλών ασθενειών κινδυνεύουν ακόμη και από θάνατο. Ο πρόεδρος διακόπτει. Κοιτάξτε, δεν είναι ερώτηση αυτό από ό,τι βλέπω στον κύριο Μαριά. Όχι, όχι, φτάνω και στην ερώτηση. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τι λέει ο κύριος Μαριάς για το θέμα αυτό αρκεί να εγκρίνουμε ψηφίσματα ή πρέπει να λάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χφαλά. Χαλα. κοιταξτε το θέμα του, Σουδάν, του Νοτιού Σουδάν είναι πάρα πολύ σοβαρά και το συζητήσαμε αυτό το οποίο κάνουμε σε αυτή τη φάση είναι να αναδείξουμε το ζήτημα και να πιέσουμε για να υπάρξουν και συγκεκριμένα μέτρα. δεν μπορούμε χωρίς συγκεκριμένα μέτρα να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. το πρώτο και βασικό είναι να πάμε στα αίτια και τα αίτια είναι η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών στο νότιο σουδάν. ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν από την κατάσταση του εμφυλίου πολέμου. όταν το δούμε αυτό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να πάρουμε μέτρα απέναντι σε αυτές τις αιτίες για να αντιμετωπίσουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεπιτή Νέκοφ. One minute. Take the floor, please. Κύριος Νέκοφ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απαγωγή χιλιάδων παιδιών τελικά είναι κάτι το απαράδεκτο ανεξάρτητα από την περιοχή του κόσμου στην οποία διεξάγεται. Ε, τέτοιες ενέργειες φυσικά χτυπούν τον πληθυσμό του Νότιου Σουδάν και η Ευρώπη θα πρέπει να προσπαθήσει να ξεπεράσει τέτοιου είδους προκλήσεις σε συνεργασία με τις διεθνείς οργανώσεις γιατί τέτοιες ενέργειες δυστυχώς γίνονται όλο και συχνότερες η κατάσταση στη χώρα αυτή είναι κρίσιμη. Τα σχολεία χρησιμοποιούνται σαν στρατόπεδα και τα παιδιά χρησιμοποιούνται σαν στρατιώτες. Ε, πάνω από 400.000 ε, παιδιά δεν πηγαίνουν πια σχολείο λόγω της κατάστασης αυτής και από ό,τι φαίνεται πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται σαν στρατιώτες η ευρωπαϊκή κοινότητα και η διεθνής κοινότητα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα μέσα που διαθέτει για να επανενταχθούν τα παιδιά αυτά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για στρατιωτικούς στόχους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εφόσον συζητήσαμε και το θέμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΙΕ, και είχα λάβει το λόγο να μιλήσω για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίω των παιδιών, πρέπει να πω ότι στο Νότιο Σουδάν, και εκεί ήθελα να αναφερθώ, βλέπουμε ότι έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς ε, τραγική παραβία, μπορεί να είναι τραγικέ παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και με φρικαλαιότητες που διαπράττονται. Εδώ πρέπει να ε, φροντίσουμε τα παιδιά που στατολογούνται και από τις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις του, ε, της συμφιλίας της σύγκρουσης και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συμφέροντα που κρύβονται πίσω από όλα αυτά ε, στο Νότιο Σουδάν και τον πλούτο του. είναι τεράστιες οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γι' αυτό την καλό να κάνω ό,τι μπορεί για να δοθεί τέρμα σε αυτά τα τραγικά συμβάντα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Καστάρντο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι πρώτη φορά που βρισκόμαστε εδώ συνάδελφοι και συζητάμε για μια άτυχη χώρα που ονομάζεται Νότιο Σουδάν. Οι πρώτες ύλε εκεί είναι μια κατάρα και δεν είναι μια ευκαιρία. Ε, δυστυχώς 10.000 παιδιά φαίνεται ότι έχουν μετατραπεί σε όργανο θανάτου ε, και αυτό δυστυχώς οφείλεται και σε εξωτερικά συμφέροντα. Εμείς ζητάμε τα παιδιά αυτά να αφαιθούν ελεύθερα, να ανοικοδομηθούν οι υποδομές της χώρας, τα σχολεία που θα επιτρέψουν την επανένταξη των παιδιών αυτών και οι ένοχοι θα πρέπει να παραπεμφθούν στην δικαιοσύνη και όλοι όσοι προσπαθούν να επωφεληθούν από το πετρέλαιο αλλά και το αίμα της συγκεκριμένης χώρας. Θα πρέπει να καταδικαστούν οι ηγέτες αυτών των ενόπλων ομάδων θα πρέπει να εγκαταληφθούν τα όπλα και να πάρουν μια σοβαρή απόφαση για την ειρήνευση της περιοχής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μιλητή. Ο κύριος Αν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αυτό ήθελα να το πω για το Ισλαμικό κράτος, αυτό ήθελα να το πω για το Σουδάν, αυτό ήθελα να το πω για τις ε, κατασχέσεις γεών στην Τανζανία. Θα πρέπει να βάλουμε και μία κίτρινη κάρτα έτσι ώστε ε, να μην μπορούν κάποιοι με την μπλε κάρτα να παίρνουν το λόγο και κάποιοι άλλοι οι οποίοι περιμένουν να πάρουν το λόγο με το Catch the Eye να μην ε, ε, έχουν την δυνατότητα να μιλήσουν ποτέ. Ευχαριστώ. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Κοιτάξτε, έχω την, την άποψη ότι ήταν σημαντικό αυτό που είπατε. Πράγματι πολλές φορές δημιουργούνται τέτοια προβλήματα, ο Επίτροπος παρόλα αυτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, το Νότιο Σουδάν ε, βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο εδώ και 15 μήνες περίπου κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε επίπεδο ανθρωπιστικών καταστροφών. Ο λόγος για την απαγωγή των παιδιών είναι πράγματι μία επιπλέον απόδειξη της πλήρους αγνόησης του ε, νόμου. Έχουν καταδικαστεί από τους διεθνείς οργανισμούς με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο. Ε, συνεχίζεται η βία εις βάρος των παιδιών από ένοπλες ομάδες, κάτι το οποίο είναι μια βασική προτεραιότητα. Εμείς συνεργαζόμαστε στενά με την εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών ε, για τα παιδιά σε περιοχές με συγκρούσεις έτσι ώστε να βρεθεί ένα τέλος. Η αντιπροσωπεία μας στην πόλη της Τζούμπα ε, προσπαθεί να συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές και να οδηγήσει τα παιδιά αυτά σε, σε ασφαλή καταφύγια και το ΕΚΟ, η υπηρεσία μας για την ανθρωπιστική βοήθεια, παρέχει έκτακτη βοήθεια έτσι ώστε να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να γλιτώσουν. Απαιτείται λοιπόν αυτό να γίνει έτσι ώστε να υπάρξει ειρήνη. Η, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει να δημοσιευθεί η έρευνα της Επιτροπής Αφρικανικής Ενότητας. Είναι μια έρευνα την οποία έχει οργανώσει η ίδια η οργάνωση αυτή και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την κατανόηση των εγκλημάτων τα οποία διαπράττονται στην Αφρικανική Ήπειρο. Εμείς θα θα λάβουμε υπόψη μας αυτά τα οποία περιλαμβάνει η έκθεση αυτή. Οι ανθρώπινες καταστροφές ε, τις οποίες βιώνουν οι πολίτες της χώρας είναι αποτέλεσμα των απαράδεκτων επιλογών των πολιτικών τους ε, ηγετών. Των πολιτικών τους ηγετών. Για μια ακόμη φορά την προηγούμενη εβδομάδα οι πλευρές αυτές αρνήθηκαν να κάνουν τις αμοιβές υποχωρήσεις οι οποίες θα οδηγούσαν σε μια συνολική ρύθμιση της σύγκρουσης. Ο πρόεδρος της Αιθιοπίας που παρεμβαίνει στην σύγκρουση αυτή ζήτησε από τις περιφερειακές αρχές να συνεχίζουν τη συνεργασία για να βρεθεί μια λύση. Εμείς θα βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κύριος Ρόντος και αυτός θα συνεχίσει τις προσπάσεις του. Έχει υπάρξει ένα ομόφωνο ψήφισμα για την επιβολή κυρώσεων εις βάρος αυτών οι οποίοι έχουν διαπράξει ε, εγκλήματα πολέμου. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να αυξηθεί η πίεση στους εμπλεκομένους χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις να πω το εξής. Έχει μεγάλη σημασία οι πλευρές που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πόλεμο να σκεφτούν λίγο και τα συμφέροντα των πολιτών της χώρας αυτής και όχι μόνο τα δικά τους συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είπαμε θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την έβρεση ταχύτατα μιας διαρκούς ειρήνης στην χώρα αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ, το, κύριε Επίτροπε. Έχω λάβει 7 σχέδια ψηφίσματος στο πέρας της συζήτησης. ολοκληρώνεται η συζήτηση. Θα γίνει ψηφοφορία εντός ολίγου.